ότι θα μετατραπεί η θανατική ποινή με μια άλλη αναλογική ποινή που θα επιβάλλεται στον καταδικαστέντα σε θάνατο. Σας ευχαριστώ κύριε Ευρωβουλευτά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει να συζητηθεί αφ' αυτού ξεχωριστά. Αυτό τελώς δεν είναι δυνατόν έτσι να ληφθεί μια απόφαση αυτοσχέδια. Οι αρμόδιες αυστριακέ αρχέ ε, με ενημέρωσαν ότι η κυρία Χέλα Ράνερ αντικαταστάθηκε από τον κύριο Χάιντ Μπέκερ από την 1η Απριλίου 2011. Θα ήθελα να καλωσορίσω το νέο συνάδελφο και να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφο 2 του κανονισμού μέχρι ότου θα έχουν ε, ε, εξεταστεί τα διαπιστευτήρια και δεν θα έχουν υπάρξει ενστάσεις. Ο κύριος Χάιντς Μπέκερ μπορεί να συνεδριάζει, να συμμετέχει συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πλήρη δικαιώματα ως Ευρωβουλευτής εφόσον θα έχει υπογράψει προηγούμενα μία γραπτή δήλωση που θα αναφέρει ότι δεν έχει κάποιο αξίωμα το οποίο είναι ασύμβατο με το αξίωμα του Ευρωβουλευτού. Βρίσκεται στην αίθουσα ο κύριος Χάιντς Μπέκερ. Σας ευχαριστώ λοιπόν εξ ονόματος όλων. Ο κύριος Τρέβο Κόλμαν. Ο κύριος Τρέβο Κόλμαν με ενημέρωσε ότι δεν είναι πλέον ε, μέλος της ομάδας ε, της Ευρώπης των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας και είναι ένας μη εγγεγραμμένος από την 25η Μαρτίου πλέον 2011. Επόμενο θέμα υπογραφή πράξεων υπό την κανονική νομική, νομοθετική διαδικασία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αποκοινούμε τον Προεδρεύμα του Συμβουλίου την Τρίτη πρόκειται να υπογραφούν τέσσερις ε, ε, δηλώσεις, τέσσερις νομικές ε, πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 74 και η, ε, τα στοιχεία αυτά είναι στη διάθεσή σας. Περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Η τελική ημερήσια διάταξη από την, στην 31η Μαρτίου υιοθετήθηκε από τη διάσκεψη των Πρόεδρων. Έχει διανεμηθεί το σχέδιο ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχουν αλλαγέ για την Δευτέρα. Για την Τρίτη όμω στη συνέχεια. Όσον αφορά την έκθεση του κυρίου Φερνάντες για τις εκτιμήσεις όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το έτος 2012 η ομάδα της Ευρώπης Ελευθεριών και Δημοκρατίας ζήτησε να αναβληθεί η ψηφοφορία για την περίοδο συνόδου του Μαΐου, του μηνός Μαΐου. Θα δώσω τον λόγο στην κυρία Αντρέασεν να υπεξηγήσει το έτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ την αναβολή της ψηφοφορίας της έκθεσης Φερνάντες από την σημερινή Ολομέλεια. Και ο λόγος είναι ξεκάθαρος και αφορούν κυρίως την παράγραφο της έκθεσης που ασχολείται με τον οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Όπου τα στοιχεία για το έργο αυτό είναι παραπλανητικά και αντιφατικά. Παράδειγμα, η αύξηση του ετήσιου κόστους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 13,5 εκατομμύρια. Το, το ποσό αυτό είναι καθυπέρβαση του αρχικού. Αρχικά είχε, προταθεί το, είχε ε, τοποθετηθεί το κόστος στα 10 εκατομμύρια και αξιωματούχος του Κοινοβουλίου με κατηγορήσει ότι λέω ψέματα, δηλώνοντας ότι οι εκτιμήσεις μου ήταν υπερβολικές. Δεν είναι τρόπος ε, αντιμετώπισης των μελών του Κοινοβουλίου αυτός. Το χειρότερο δε πρόεδρε είναι ε, το, η σαφή σύγκρουση ε, συμφερόντων όταν ε, η πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του οίκου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας έστω και χωρίς αμοιβή. Σε καμία ένα άλλο κοινοβούλιο δεν θα ήταν δεκτό τέτοια σύγκρουση συμφερόντων. Ευχαριστώ, διακόπτει ο πρόεδρος. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί και μέχρι να ξεκαθαριστεί η ψηφοφορία δεν πρέπει να συνεχιστεί. Θα ήθελα να ξέρω, υπάρχει κάποιος που υποστηρίζει το αίτημα, που θέλει να υποστηρίξει το αίτημα. Κύριε Σπερόνια. Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι σκόπιμη η αναβολή αυτή τέσσερις πέντε εβδομάδες είναι απλά για να εξεταστεί διεξοδικότερα ένα ζήτημα που όπως ακούσαμε μόλις περιλαμβάνει την χρηματοδότηση εκατομμυρίων ευρώ από, πλευρά, από τις τσέπες των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Εγώ ζητώ λοιπόν την υπερψήφιση της αναβολής. Υπάρχει κάποιος που θέλει να λάβει θέση κατά. Ο κύριος Λαμασούρ καταρχήν. Πρόεδρε, να πω δύο πράγματα. Πρώτον, η Επιτροπή Προπολογισμών έκανε τη δουλειά της και έθεσε το σχέδιο των estimates, των εκτιμήσεων του προπολογισμού του Κοινοβουλίου στο 2012 σε θέση εξέταση, συζήτηση και ψηφοφορία από το Κοινοβούλιο, από την Ορομέλεια. Σύμφωνα με τις διαδικασίες και σύμφωνα με ό,τι είχαμε κάνει και πέρυσι. Υπάρχουν διστάμενε απόψεις μεταξύ των ομάδων μπορούν να εκφραστούν. Δεύτερον, δεν θέλω να δηλώνει η κυρία Αντρέασεν που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμών, μέλος του Συμβουλίου Προσανατολισμού του οίκου Ευρωπαϊκής Ιστορίας, έχω προσωπικά πρόβλημα σύγκρουσης συμφερόντων. Δεν είμαι εκεί προσωπικά, αλλά ως πρόεδρο τη επιτροπή Προπολογισμών που ορίστηκε από την Επιτροπή Προπολογισμών για να την προσωπεύω στο όργανο αυτό. Με τον ίδιο τρόπο που ο πρόεδρο τη επιτροπή Πολιτισμικών Υποθέσεων εκπροσωπεί την Επιτροπή αυτή στο ίδιο όργανο. Φυσικά διακόπτεται. Αν κάποιο το αμφισβητεί είμαι έτοιμο να θέσω την εντολή μου στη διάθεση του σώματο, αλλά δεν μπορώ να ακούω εκφράσει όπω σύγκρουση συμφερόντων κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να προσέχουμε πώς να μην προσβάλλουμε τον κόσμο. Ευχαριστώ. vote. Θα ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ του αιτήματο της κυρίας Ανδρέασεν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το αίτημα. Τετάρτη. Συζήτηση για την εσωτερική αγορά. Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ζήτησε να μπορούν να υποβληθούν αιτήματα ψηφίσματος για να, συζητηθεί, για να αντιμετωπιστεί το, συζήτηση, το θέμα συζήτησης δημοσίων ε, συμβάσεων. Είναι προτάσεις ψηφίσματος. Κάποιος από την ομάδα ΕΛΚ θα μπορούσε να παρουσιάσει το σημείο αυτό. Ποιος θα παρουσιάσει το αίτημα αυτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η ομάδα του ΕΛΚΑ για την νομοδότηση του Επιτρόπου ε, Μπαρνιέ για τι δημόσιε προμήθειε και τη μεταξέλιξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέλει να συμπληρώσει με μια γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό θα ολοκλήρωνε και θα έδινε νόημα. Γι' αυτό ζητούμε υποστήριξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάποιο θέλει να λάβει το λόγο για να μιλήσει κατά τη προτάσεω. Κύριε Μπερές. Όχι. Κύριε Κυρία Γκέπχαρτ. Παρακαλώ. Γκέπχαρτ, όχι Μπερές. Υποστηρίζω όμω την πρόταση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Είναι απόλυτα λογικό να συζητηθεί το θέμα αυτό. Απλώς θα ήθελα να παρακαλέσω, και το έχουμε συζητήσει και με τον συντονιστή, τον κύριο Σφαπ, αυτή την εβδομάδα να μην, να μην ψηφίσουμε το ίδιο το ψήφισμα, να αφήσουμε την ψηφοφορία για το Μάιο, γιατί δεν είχαμε προλάβει μεταξύ μα οι ομάδε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Άρα ναι, υπέρ τη εγγραφή στην ημερήσια διάταξη, ναι, υπέρ του ψηφίσματο, αλλά παρακαλούμε η ψηφοφορία να γίνει το Μάιο μόνο. Καλώς Ευχαριστώ. Ποιο θέλει να μιλήσει κατά τη πρόταση αυτή. Κατά. Δεν βλέπω κάποιον να θέλει να λάβει το λόγο. Ποιοι είναι υπέρ της προτάσεως του ΕΛΚ κατά αποχές εγκρίνεται το αίτημα. Προθεσμίες για το, το σημείο αυτό είναι οι εξής. Προτάσεις ψηφισμάτων, προθεσμία, αύριο στις 10 το πρωί. Τροπο, τροπολογίες και κοινά ψηφίσματα, κοινές προτάσεις ψηφίσματος, Τετάρτη, μεθαύριο, 10 η ώρα το πρωί. Τροποποιήσει στα κοινά, στις κοινέ προτάσεις ψηφισμάτων, Τετάρτη, μεθαύριο, την ίδια μέρα δηλαδή, 11 το πρωί. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την 5η, 7 Απριλίου, στις 12. Πολύ περιορισμένο το χρονικό διάστημα. Για την 5η τώρα η ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών στην Ευρώπη ζήτησε να γίνει συζήτηση για το θέμα του Ai Weiwei στην Κίνα, ζητώντας να συμπεριληφθεί το θέμα αυτό στις συζητήσεις βάσει του άρθρου 122 του κανονισμού την 5ο απόγευμα, αντί της αρχικά σα συζήτησης για τη Ζιμπάμπουε. Κύριε Φερχόφστατ, έχετε ζητήσει το λόγο για να υποστήριξετε τη θέση αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Άι Βέι είναι ο πιο γνωστός καλλιτέχνης και αντιφρονών Κινέζος και είχε πάντα τη δυνατότητα να εκφράζεται ελεύθερα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Πεκίνου την Κυριακή και μάλλον είναι φυλακισμένος. Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή όχι μόνο για να διαμαρτυρηθούμε για την κράτησή του από τις Κινέζικες Αρχές, θα ήθελα να πω ότι θα έπρεπε να επαεξετάσουμε τη συμμετοχή μας στην δεύτερη σύνοδο κορυφής Ευρώπης, ηγετών ε, Ευρώπης-Κίνας στην, ε, τον άλλο μήνα, στο Πεκίνο. Πιστεύω ωστόσο ότι είναι αναγκαίο να γίνει ένα επίγον ψήφισμα για το θέμα αυτό όσο πιο γρήγορα γίνεται, ούτως ώστε να αυξηθεί η πίεση προς τις κινησικές αρχές για την απελευθέρωση του κ. Άι Βέι. Αρχικά είχαμε σκεφτεί την Πέμπτη να αντικαταστήσουμε το ψήφισμα για την Ζιμπάμπουε με την κράτηση του IVV. Μετά από μια συζήτηση σύντομη, πρόεδρε, μπορεί να βρούμε μια καλύτερη λύση. Να θέσουμε Τετάρτη το θέμα της ακτής ελεφαντοστού και το κενό που θα απελευθερωθεί την Πέμπτη να μπει το ψήφισμα για τον IVV. Μίλησα με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες, συμφώνησαν με την διαμόρφωση αυτή της ημερήσιας διάταξης. Βεβαίως, είναι περίπλοκο το να γίνει μια τέτοια αλλαγή. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε επακριβώς τη διαδικασία. Αυτό σημαίνει, πρώτα απ' όλα, ότι πρέπει να υπάρξει πρόταση για αλλαγή θέση στο θέμα της ε, ακτή του Ελεφαντοστού. Από πέμπτη απόγευμα δηλαδή ακτή του Ελεφαντοστού να συντηρηθεί την ε, Τετάρτη, μάλλον στις 8. Γιατί δεν βλέπω αλλού περιθώριο. Μισή ώρα με 45 λεπτά στις 8 το απόγευμα για τη Ζιμπάμπουε και έτσι μας περισσεύει ο, χώρος, ο χρόνος για τον Ai για να του προσφέρουμε αυτή τη βοήθεια. Συμφωνούμε όλοι. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Θέλει κανείς να τοποθετηθεί υπέρ ή κατά της προτάσεως. Ε, υπέρ παρακαλώ. Υπέρ της προτάσεως. Ας ψηφίσουμε τότε. Ο κύριος Φόμποτα. Πρόεδρε, πολύ σύντομα υπέρ. Είναι τόσο πυκνή όμως η μερίση διάταξη Τετάρτης. Γι' αυτό θα παρακαλούσα και το Συμβούλιο και η Επιτροπή να περιοριστούν όσο δυνατόν πιο σύντομες ομιλίες στις παρεμβάσεις τους και να είναι πολύ προσεκτική με το χρόνο, ιδιαίτερα και την Αντιπρόεδρο που είναι εδώ. Παρακαλώ λοιπόν να μα υποστηρίξετε και εσεί βέβαια μέσω των Αντιπροέδρων στην, τήρηση, στην όσο δυνατόν ε, αυστηρή τήρηση του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο, το αναφέρω και στο Προεδρείο. Ποιο υποστηρίζει την πρόταση αυτή για να κατά. Ευχαριστώ. Άρα λοιπόν το θέμα του Άιουεϊ στην ε, Κίνα θα συζητηθεί την Πέμπτη το απόγευμα. Η δε ακτή του ελεφαντοστού περίπου στις 8 το βράδυ την Τετάρτη. Άλλο ένα θέμα, μια πρόταση της κυρίας Γκέπχαρτ. Όχι. suggested we take the vote in May, not in April. And we didn't. Decision, colleagues. Είναι η τελευταία απόφαση που έχουμε να λάβουμε για την ημερήσια διάταξη. Κυρία Γκέπχαρτ, θα παρακαλέσω για άλλη μια φορά να επαναλάβετε την πρότασή σα, να διατυπώσετε την πρότασή σα. Κύριε Πρόεδρε, παρακάλεσα η ψηφοφορία για το ψήφισμα το σχετικό με τις δημόσιες προμήθειες να μετατεθεί στο Μάιο, στην Ολομέλεια του Μαΐου. Άρα οι προθεσμίες για την κατάθεση των ε, ψηφισμάτων και των τροπολογιών τους μπορεί αντίστοιχα να αναβληθεί. Ευχαριστώ, λέει ο Θέλει κανείς να λάβει το λόγο υπέρ της προτάσεως αυτής, κατά κάποιες παρατηρήσεις. Δεν βλέπω να είναι καν... Ο κύριος Περόνι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεδομένης της... Δεδομένου του θέματος και του χρόνου που έχουμε για να υποβάλουμε τροπολογίες θεωρώ ότι είναι επαρκή ο χρόνο και δεν νομίζω ότι αρκεί, ε, χρειάζεται να υποστηρίξουμε την πρόταση αυτή. Ποιο υποστηρίζει την πρόταση, κυρία Γκέπχαρτ, παρακαλώ, παρακαλώ, σηκώστε το χέρι υπέρ της προτάσεως. Κατά τώρα. Ευχαριστώ. Εντάξει, λοιπόν, η πρόταση σας γίνεται δεκτή, κυρία Κεπχάρτ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα, εφόσον προσδιορίστηκε η οριστική μερίσια διάταξη, μπορούμε να προχωρήσουμε στο πρώτο μας θέμα, που είναι η έκθεση της κυρίας Γκίομ, η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της διεθνούς προστασίας στα κράτη-μέλη. Η κυρία Νετφέλτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Δεν ε, ήξερα και σε ποιο σημείο τη ημερήσια διάταξη να ζητήσω το λόγο. Πριν από δύο εβδομάδες, πριν από μια εβδομάδα περίπου, η διοίκηση του Κοινοβουλίου ε, λόγω κάποιων κυβερνοαπειλών απεφάσισε να κλείσει το διαδίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για μια ολόκληρη εβδομάδα. Δεν καταλαβαίνω πώ είναι δυνατόν να λαμβάνονται τι αποφάσει και να αποστερούμαστε την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μα ταχυδρομείο για μια ολόκληρη εβδομάδα. Θα ήθελα να ενημερωθώ λοιπόν πόσο σοβαρό ήταν ο κίνδυνο, αν ήταν μόνο προληπτικό το μέτρο και σε τελευταία ανάλυση πόσο ευάλωτο είναι το ηλεκτρονικό μα σύστημα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Θα το επαληθεύσουμε και θα σα ενημερώσουμε.